Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 19 Απριλίου βάσει του άρθρου 149 έχει μοιραστεί. Την Τετάρτη το ΕΛΚ ζήτησε να προσθεθεί ω τέταρτο σημείο στη σημερινή ημερήσια διάταξη δήλωση τη ε, Αντιπροέδρου Εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ε, η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί με ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Θέλει κάποιο να υπερασπιστεί την ε, πρόβλεψη του θέματο αυτού, ο κ. Γκονσάλε Πρόεδρε, όταν δώσαμε το βραβείο Ζαχάροφ στην αντιπολίτευση τη Βενεζουέλα, εμεί εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναλάβαμε κάποια δέσμευση απέναντι στη Βενεζουέλα. Στις 20 Μαΐου στη Βενεζουέλα θα γίνουν κάποιες ψευτοεκλογές και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να μην λάβουν χώρα. Γι' αυτό η καλύτερη βοήθεια που θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε είναι να εγκρίνουμε ψήφισμα που θα λέει τα εξή. Πρώτον, ότι δεν θα αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα τέτοιων ψευδοεκλογών. Δεύτερον, ότι ζητάμε από το καθεστώ του Μαδούρο να μην προβεί στι εκλογέ αυτέ, αλλά να μπει σε διάλογο με την αντιπολίτευση. Και τρίτον, να μην συμμετέχουμε σε διεθνή παρατήρηση των εκλογών αυτών, γιατί τότε θα ήταν σαν ήμασταν συνένοχοι του Μαδούρο. Ο Μαδούρο εκλέχτηκε σε εκλογές που αναγνώρισαν όλοι. Αλλά τώρα, αν ξαναβγεί, δεν θα έχει νομιμότητα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να στηρίξουμε την βενεζουαλινή αντιπολίτευση όπως δηλώνει και το βραβείο Ζαχάροφ που τους ε, αποδώσαμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Κόζο Περμούη που έχει να προβάλλει αντίρρηση. Εμείς είμαστε κατά της πρότασης αυτής γιατί είναι ακατάλληλη με το ζόρι και η μόνη πρόθεση που έχει είναι να παρεύει να αναμειχθεί σε κάποιες εκλογές που ξέρετε ότι δεν θα κερδίσουν οι φίλοι σας το Λαϊκό Κόμμα το παραδέχεται. Οι εκλογές των φίλοντας με το ίδιο εκλογικό συμβούλιο ενέκρινε τις εκλογές της συνέλευσης. Κέρδισαν οι φίλοι σας τότε και δεν είχατε πρόβλημα, αλλά με το ίδιο εκλογικό συμβούλιο τώρα καταγγέλλετε τις επόμενες εκλογές γιατί δεν είναι υποψήφιοι δικοί σας. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν ε, γίνεται τέτοιο πράγμα. Εσείς λοιπόν θέλετε ε, αστάθεια στην χώρα και να πετύχουν οι φίλοι σας με την βία στους δρόμους. Σταματήστε να ενισχύετε το χάος και βοηθήστε στην κανονικότατα στη χώρα. Πείστε τους φιλαράκους σας εκεί να συνομιλήσουν και να μπουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Η κυρία Ευχαριστώ. Η κατάσταση στην Βενεσουέλα είναι πολύ σοβαρή και γι' αυτό και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μεγάλη σοβαρότητα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 156 το αίτημα του ΕΛΚ, γιατί αναφέρεται εκεί ότι δεν μπορεί, ε, εάν δεν έχει κατατεθεί 24 ώρες νωρίτερα το αίτημα εκ Προ του βουλευτέ, δεν μπορεί να ψηφιστεί. Πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί. Και βέβαια υπάρχει η εξαίρεση των όλων ε, κατεπηγόντων, ε, κατεπηγόντων κατεπηγουσών καταστάσεων. Εδώ έχουμε μια κατάσταση που γνωρίζουμε εδώ και δύο μήνε, άρα κατεπήγουσα δεν είναι. Και άρα θα πρέπει όλε οι ομάδε και όλοι οι βουλευτέ να έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν το κείμενο, να προβάλλουν τι αντιρρήσει του. Δεν μπορεί μόνο μεγάλε ομάδε με τον πρόεδρο να αλλάζουν του κανόνε, Κατά το δοκούν υπάρχουν οι κανόνε και πρέπει να εφαρμόζονται. Κύριε Κονζάλες Μόνς. Εάν η δημοκρατία στη Βενεζουέλα είναι κάτι σημαντικό, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να μην αγωνιζόμαστε για αυτήν για διαδικαστικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν η διαδικασία να είναι πιο σημαντική από τη δημοκρατία. Όταν η διαδικασία μπαίνει πάνω από τη δημοκρατία, αυτό αποτελεί άλοθη και μόνο για να μην στηρίξουμε τη δημοκρατία. Συνεπώς, το κατεπήγον, διακόπτει ο μιλητής, το επίγον δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε. Είναι σαφέ. Είναι στο χρονοδιάγραμμα. 20 Μαου θα γίνουν οι εκλογέ. Δεν έχουμε στο μεταξύ άλλη ολομέλεια για να μπορέσουμε να αποφανθούμε. Λοιπόν, ή θα αποφανθούμε τώρα, ή αλλιώ δεν θα υπάρξει ψήφισμα από την πλευρά μα. Και εγώ προτιμάω να υπάρξει ψήφισμα. Εσύ μπορεί να προτιμάτε να μην υπάρξει ψήφισμα. Ε, για ένα ενδιάμεσο ψήφισμα, δεν ξέρω. Να έχουμε συζήτηση και αυτό που έχει υποστηρίξει σε διάφορα ψηφίσματά του το Κοινοβούλιο νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί από μία δήλωση του Προέδρου εκ μέρους όλων μας. Κύριε Γκονζάλες Πόντς. Κύριε Γκονζάλες Πόντς. Κύριε Γκονζάλες Πόντς, por favor. Αντιλαμβάνομαι ότι ζητάτε συζήτηση χωρίς ψήφισμα μετά από αυτά που είπε η κυρία Κέλλερ. Και μετά ζητάτε δήλωση του Πρόεδρου, έτσι, που να συνοψίζει ουσιαστικά το κείμενο του ψηφίσματος που έχει ψηφιστεί στο μεταξύ εδώ. Αυτό ζητάτε. Αυτή είναι μια συνενετική πρόταση. Αν δεχτείτε αυτή την πρόταση, εντάξει, μας κάνει. Αλλιώς θέλουμε να ψηφίσουμε την πρότασή μας. Μια ναι, Κέλλερ. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογισμό αυτό, γιατί οι προηγούμενα ψηφίσματα που έχουμε εγκρίνει δεν λέγαν τίποτα για το ψηφίσματα του Μαΐου. Θα έπρεπε νωρίτερα να το έχετε ζητήσει Δύο μήνες τώρα, όπως είπα, και αν θέλετε για δίποτε δήλωση, ε, πώς είναι δυνατόν να εγκριθεί μια δήλωση την οποία μόνο μια ομάδα έχει εγκρίνει και που δεν έχουν παρακολουθήσει οι άλλοι σε κανένα κομμάτι της διαδικασίας. Δεν το επιτρέπει το άρθρο 156. Κυρία Κέλλερ, υπάρχει πρόταση του κυρίου Γκονζάλης Πόνς να γίνει συζήτηση χωρίς ψήφισμα με δήλωση του Προέδρου. Σε συμφωνία με το προσφατότερο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο. Συμφωνείτε ή να ψηφίσουμε. Βεβαίως. Πάντα μπορείτε να επαναλαμβάνετε αυτά τα οποία έχουμε πάλι σε ένα ψήφισμα. Αλλά το προηγούμενο ψήφισμα δεν αναφέρει τίποτα για εκλογές του Μαΐου και ως εκ τούτου πρέπει να ψηφίσουμε. Ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ο κύριος Κονσάλες Πώς προκειμένου να υπάρχει συζήτηση με ψήφισμα μαζί ζητεί να γίνει κατεπίγουσα η συζήτηση αυτή. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ψήφισμα. Η κυρία Κέλλερ όμως λέει ότι η Δάλος, εάν δεν ζητηθεί το κατεπήγον, δεν είναι δυνατόν και νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Κέλλερ δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με ψήφισμα, χωρίς να ζητηθεί το κατεπήγον. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε αν η Ολομέλεια θέλει συζήτηση κατεπήγοντος για το θέμα αυτό. Με ψήφισμα. Εάν αυτό το αίτημα δεν περάσει, τότε περνούμε σε συζήτηση χωρίς ψήφισμα. Ψηφίζουμε λοιπόν. Εάν θέλουμε συζήτηση κατεπήγοντος για ψήφισμα στην υπόθεση της Βενεζουέλας και ξεκινάει η ψηφοφορία. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Η πρόταση γίνεται δεκτή, συζήτηση με ψήφισμα. Και ως εκ τούτου το θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και μετά το ψήφισμα θα δεθεί ψηφοφορία την 5η. 2 Μαΐου ένα λεπτό, αγαπητοί συνάδελφε. Έχει γίνει η συζήτηση. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και μετά εσείς θα λάβετε το λόγο. Περιμένετε μόνο. δεν τηρείται τον κανονισμό. Γιατί για ένα ψήφισμα οι ομάδες πρέπει να έχουμε στη γλώσσα μας το ψήφισμα αυτό τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Μη στρεβλώνετε τον νόμο όπως κάνει το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία για να καλύψει τη διαφθορά. Μη στρεβλώνετε τον νόμο. Εάν δεν πρόκειται για συζήτηση κατεπήγοντος, επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο ήδη είπε με πολύ απλό και σαφή τρόπο η κυρία Κέλλερ. Έδωσα δίκαιο λοιπόν στην κυρία Κέλλερ σε σχέση με το θέμα του αν θα γίνει συζήτηση. Ωστόσο, ο κύριος Κονσάλες Πόν ζήτησε κατεπήγουσα συζήτηση. Η κατεπήγουσα συζήτηση επιτρέπει την έγκριση, διατύπωση και έγκριση ψηφίσματος. Άρα, μέχρι τις 6 θα γίνει η καταθέση της των προτάσεων ψηφισμάτων. Δευτέρα, ε, Τετάρτη 2 Μαΐου, τροπολογίες μέχρι τις 9 ε, το βράδυ, προτάσεις χωριστών ψηφισμάτων Τετάρτη μέχρι τις 11 το βράδυ, Τετάρτη 2 Μαΐου δηλαδή σήμερα, μέχρι τις 11 το βράδυ, ψηφοφορία την Πέμπτη. Η ομάδα της ΓΚΟΕ έχει ζητήσει μετά ε, την ε, συζήτηση μια, ε, μια δήλωση από το Συμβούλιο για την εφαρμογή από την Ισπανία των διεθνών διατάξεων σε σχέση με την σεξουαλική γενετήσια βία στην υπόθεση Μανάντα. Παρακαλώ τον κύριο Πένιας να παρουσιάσει το αίτημα της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ. Κυρία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πολλές Ισπανίδες νιώθουν ότι δεν τις προστατεύουν οι αρχές. Πριν από μία εβδομάδα στην Αβάρα είχαμε μια δίκη και αποφάσισε η αθώση μετά από έναν πολλαπλό βιασμό. Πέντε άνθρωποι που ονομάζονται Λαμανάδα οι ίδιοι πρέβησαν σε βιασμό και σε και η απόφαση λέει ότι δεν πρόκειται για βιασμό, ότι πρόκειται για μία απλώς ε, βία γιατί δεν υπήρξε ολοκλήρωση. Είναι βάρβαρα όλα αυτά. Η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μιλάει για τον βιασμό ότι είναι κάθε σεξουαλική πράξη στην οποία δεν συνενεί το θύμα. Έξι ευρωπαϊκές χώρες όμως έχουν δεχτεί αυτό τον ορισμό του βιασμού. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο. Προκειμένου αυτή η κοινωνική μάστιγα να μην επεκταθεί περισσότερο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να γίνει αυτή η συζήτηση για να αναγνωρίσουμε τι σημαίνει διασμός και να υπάρχει ένας ορισμός ο ίδιος για όλες τις χώρες, ώστε να μην επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ. Κυρία Φεραγκούτ, παρακαλώ, για να αντικρούσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε και εμείς με την οργή και την αγανάκτηση, γιατί θέλουμε μηδέν ανοχή σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάτι τέτοιο είναι και η σεξουαλική βία. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης όντως πρέπει να τηρείται από όλες τις χώρες επικρίσεις ε, πάντως σε δικαστικές ε, αρχές είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε γιατί οι δικαστές αποφασίζουν σε μια δημοκρατία σύμφωνα με τον νόμο. Οπότε δεν μπορούμε να δικάσουμε ένα δικαστή για την απόφασή του. Αλλιώς υπάρχουν τα δικαστικά μέσα που προβλέπονται στο ποινικό δίκαιο. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει, να πάει υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο κτλ. Οπότε, ναι, να γίνει συζήτηση. Ναι, να συζητήσουμε μελλοντικέ αλλαγές προκειμένου να ε, συνυπογράψουμε όλη τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά υπάρχει διάκριση εξουσιών. Άλλο νομοθετική εξουσία, άλλο δικαστική εξουσία, οπότε μην τα μπερδεύουμε αυτά. Δεν θα κάνουμε καθόλου καλό στους πολίτες. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Όχι, με εντάξει, λέει η κυρία Κέλλερ. Ψηφίζουμε την πρόταση της ομάδας Γκουέντζιελ, Παρακαλώ, ζητάτε το λόγο. Με ηρεμία, παρακαλώ. Με ηρεμία. Ονομαστικά ψηφίζουμε την πρόταση της ομάδας GUE NGL άρχεται η ψηφοφορία. Il Εγκρίνεται η πρόταση. Επομένως, ζητείτε δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής για την εφαρμογή από πλευρά τη Ισπανία των διεθνών προδιαγραφών και αρχών σε σχέση με την γενετήσια βία εν ώψη προς, της πρόσφατης υπόθεσης Λαμανάντα και σε σχέση με την Σύμβαση για την Προστασία των Θυμάτων. Η ομάδα των Πρασίνων Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία έχει ζητήσει την εμμυρίση διάταξη να συμπεριληφθεί συζήτηση με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον για τους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ε, χάλιβα και το αλουμίνιο και απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Σκακέλερ για να εξηγήσει το αίτημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι δασμοί που μπορεί να επιβληθούν ή όχι από τι ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εμείς ως συνονομοθέτες παραμένουμε στο σκοτάδι σε σχέση με τα όσα αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα σήμερα κάποιοι συνάδελφοι τη Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είχαν μια κάποια ενημέρωση, αλλά αυτή την ενημέρωση πρέπει να ε, την γνωρίζουν και όλοι οι βουλευτέ, αλλά και το ευρύ κοινό. Ε, για το τι μπορεί να επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω μάλιστα με τη μορφή μια νέα εντολή για νέε διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ μέχρι και το τέλο του μήνα. Ακόμα εμεί στο Κοινοβούλιο πρέπει να γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει αυτή η εντολή και τι θα διαπραγματευτεί ή τι δεν θα πρέπει να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν είναι να το γνωρίζουμε, πρέπει να το συστήσουμε σήμερα στην τρέχουσα σύνοδο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τη σύνοδο τη δεύτερη του Στρασβούργου, γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Γι' αυτό σα καλώ να συμφωνήσετε σε μια συζήτηση για την τρέχουσα μήνυ ολομέλεια για το θέμα αυτό, ώστε να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να εκφέρει γνώμη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ για να αντικρούσετε. Κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ συχνά στην πολιτική κάποιοι μιλάνε ταχύτερα από ό,τι σκέφτονται. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, λοιπόν, καλό το σώμα να μην δεχθεί αυτή την ε, συζήτηση με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρέχουσα μήνυ Ολομέλεια. Πολύ ευχαριστώ, βέβαια, να το συζητήσουμε. Όχι ότι θεωρώ ότι ε, ε, έχουμε πολύ αποκλίνουσες απόψεις σε σχέση με τους δασμούς που θέλει να επιβάλλει στο Χάλιβα ο Τραμπ. Είναι παράνομοι. Αλλά όλα αυτά ανακοινώθηκαν μόλις χθε, ούτε καν τις λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε ούτε καν τι λεπτομέρειε τη ίδια για την επιβολή δασμών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και να διαβάσουμε και να αναλογιστούμε καλύτερα πριν τι έχουμε να πούμε πριν να το πούμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε και καμιά άλλη ευκαιρία. Έπεται μια δεύτερη ολομέλεια στο τέλο Μαΐου. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να συλλέξουμε όλο το υλικό, όλε τι λεπτομέρειε και να διατυπώσουμε το σαφέ και περίφραστο μήνυμα του Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει πριν να γνωρίζουμε ακριβώ τι έχουν αποφασίσει από τη Ουάσιγκτον ο Πρόεδρος. Για μένα προσωπικά είναι απαραίτητο να σημειώσω ότι η κυρία Σκακέλερ πάντοτε σκέφτεται προσεκτικά πριν να μιλήσει. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ε, δεν τυπώνεται τέτοιο ισχυρισμό πω μιλάει χωρί να σκέφτεται. Αλλά περνώ τώρα στην ονομαστική ψηφοφορία υπέρ τη προτάσεω των Πρασίνων με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το αίτημα απερίφθη. 'Την ε, Πέμπτη έχει προσθεθεί ακόμη ένα σημείο, το θέμα της γενετικά του γενικά, γενετικά τροποποιημένου ζαχαρότευτλου 7 Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνεται, συμπεριλαμβάνεται στην μερίσια διάταξη και έτσι ορίζεται και η μερίσια διάταξη τη τρέχουσα συνόδου και περνώ στις δηλώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόφαση της δέσμης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Γιουνκέρ που δέχτηκε να έρθει να παρουσιάσει την πρόταση για το νέο δημοσιονομικό